και θα σας ρωτούν στην αρχή της επόμενης Συνόδου Ολομέλειας. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους αποδέκτες που αναφέρονται σε αυτά. Σας ευχαριστώ.